Pan Przewodniczący! E, proszę Κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται οι εργασίε της Ολομέλειας. Τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης είναι στη διάθεσή σας. Έχετε κάποια σχόλια ή ερωτήσεις. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι εγκρίνονται τα πρακτικά αυτά. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι ο γύρος ερωτήσεων με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για αλληλοδιάδοχη ευκαιρία σειρά έχουμε αυτή την ευκαιρία να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Υπενθυμίζω τους κανόνες. Ένα λεπτό για την ερώτηση, ένα λεπτό για την απάντηση μπορεί να υπάρξουν και ένα, μια επερώτηση σε μισό λεπτό με απάντηση μισού λεπτού επί οποιοδήποτε θέματος εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων θα ακολουθήσει μετά το δεύτερο τμήμα της συνεδρίασής μας για τα επόμενα 30 λεπτά θα κάνουμε λόγο για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ζητήσουμε θα δοθεί δυνατότητα στους ευρωβουλευτές να διατυπώσουν ερωτήσεις με την ίδια διαδικασία. Ένα λεπτό για τις ερωτήσεις και ένα λεπτό για την απάντηση του κυρίου Μπαρόσο. Η πρώτη ερώτηση από τον εκπρόσωπο του ΕΛΚ, τον κύριο Ότμαρ Κάρας. Παρακαλώ κύριε Αντιπρόεδρε Ότμαρ Κάρας. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Το Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών, η Ελλάδα, η Στρατηγική 2020 ψάχνουμε για απαντήσεις για την οικονομική, χρηματοοικονομική κρίση και για τα αναγκαία μέτρα <clears throat> πολύ γοργά φτάνουμε στα όρια των δυνατοτήτων των σημερινών συνθήκων και από την άλλη πλευρά όμως κάποια κράτη-μέλη αντί να στρέψουν το βλέμμα προς την Ευρώπη έχουν μια εθνικιστική τάση, προστατευτική τάση και διακυβερνητική πολιτική τάση. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα, να δημιουργηθούν οι αναγκαίοι κοινοτικοί στόχοι που θα καθοριστούν και να υπάρξουν αξιόπιστα ευρωπαϊκά μέσα τα οποία θα δημιουργήσουμε για να χρησιμοποιήσουμε για να είμαστε αποτελεσματικοί και να βρούμε τι σωστέ αποτελεσματικέ απαντήσει. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχετε τον λόγο, Πρόεδρε της Επιτροπής, για να απαντήσετε. Δεν είναι, ε, πρέπει να μας εκπλήσει. Υπάρχουν ε, κάποιοι πολιτικοί που κάνουν μια δική τους, δίνουν μια δική τους ερμηνεία στη συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Η συνθήκη της Λισαβόνας θέλει ακριβώς να ενισχύσει την ευρωπαϊκή διάσταση, τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την λήψη αποφάσεων με ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία και τον αυξημένο ρόλο της χρηματοοικονομικής εποπτείας στα οικονομικά θέματα. Είναι όμως ε, κάτι το οποίο συμβαίνει παρόλα αυτά. Φυσικά σε σχέση με την Επιτροπή όπως είμαστε θέματοφύλακα της ε, συνθήκης σύμφωνα με το άρθρο 17 της συνθήκης της Λισαβόνας έχουμε καθήκον να προστατέψουμε το ευρωπαϊκό δίκαιο και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα στέναροι προστατεύοντας ε, το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο αλλά επίσης να προαγάγουμε πρωτοβουλίες, να αναλάβουμε τον ηγετικό ρόλο για αυτές τις πρωτοβουλίες. Θα κάνουμε τη δουλειά μας υποβάλλοντας από πλευράς μας προτάσεις που ελπίζω θα υποστηριχθούν από την Ευρωβουλή. Στι πολιτικέ μου κατευθυντήριε γραμμέ αναφέρω μια ειδική, την ειδική σχέση με την Ευρωβουλή και θέλω αυτή να γίνει πραγματικότητα. Σα ευχαριστώ. Εσεί έχετε τον λόγο για υπερώτηση, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, στη Μαδρίτη ο επίτροπο Όλι Ρέ ένα πακέτο πρότεινε το οποίο δεν έχει ακόμα εγκριθεί αλλά με κυρώσεις <clears throat> για την συζήτηση για να υπάρξουν δυνατότητες κυρώσεων Τώρα, σε σχέση με τις ε, κυρώσεις, ε, σε σχέση με τα κράτη-μέλη, θα ήταν η λάθος ε, προσέγγιση. Αντίθετα, οι κοινοί στόχοι, οι κοινοί, τα κοινά προγράμματα και σχέδια, τα κοινά μέσα εργαλεία πρέπει να καθοριστούν, τα οποία χρειαζόμαστε και μόνο τότε, όταν θα έχει γίνει αυτό, τότε να κάνουμε λόγο για κυρώσεις, όταν δεν θα υπάρχει αλληλέγγυα συμπεριφορά από πλευρά των κρατών, για να μπορέσουμε να θέσουμε κέντρα βάρους που πρέπει να ακολουθηθούν. Ευχαριστώ. Όπως είπα κύριε Καράσα, δεν υπάρχει κάποια, προ... κάποια ηλυμένη απόφαση. Μια πρώτη συζήτηση έγινε με του Υπουργού Οικονομικών και θα υποβάλει την ανακοίνωσή τη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον επόμενο μήνα για την ενισχυμένη ε, χρηματοοικονομική διακυβέρνηση και να μπορέσουμε να ε, οδηγηθούμε στη σωστή ισορροπία για το Σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη ώστε να υπάρξουν οι αναγκαίε δράσει μακροοικονομικά στι ευρωπαϊκέ πολιτικέ και θα δούμε την δυνατότητα δημιουργία ενό μηχανισμού αντιμετώπιση. Ε, θα επικεντρωθούμε όμω στην ίδια την ουσία. Πιστεύω ότι είναι δυνατόν με, αυτή, με το σημερινό πλαίσιο των συνθήκων να καταφέρουμε πολλά περισσότερα όσον αφορά την ευθυγράμμιση των κρατών μελών σε σχέση με τα οικονομικά. Αν υπάρχει η βούληση των κρατών μελών να συνεργαστούν και να σεβαστούν τι συνθήκε. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και τώρα εξ ονόματο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ο πρόεδρο κύριο Μάρτιν Σούλτ. Σα ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, το άρθρο 125 της Συνθήκης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει την bailout clause, την ρήτρα, να, την απαγόρευση να υπομίζονται κάποια, τα κράτη-μέλη τα χρέη των άλλων κρατών. Πώ ε, τοποθετήστε στο πακέτο για την Ελλάδα που τώρα οδηγεί στο ότι χώρες όπως η Ομοσπονδιακή Γερμανία χρήματα για τρία χρόνια με 5% θα δανείσουν οι Γερμανοί στο, ε, στην Ελλάδα που με μια δέσμευση τριετή σε κατά 1,5% θα υπάρξει άφηση και έτσι 4,5 δις θα είχαμε 26 εκατομμύρια κέρδος από πλευράς ε, τους. Δεν λέει η bailout clause ότι αν δεν επιτρέπεται τα χρέη ενός κράτους να τα αναλάβει ένα άλλο κράτος ότι δεν μπορεί να αποκομίζει κέρδη ένα κράτος ε, λόγω του χρέους ενός άλλου κράτους είσαστε πρόθυμος ε, να δεχθείτε αυτό τον απαράδεκτο μηχανισμό. Απόλυτα απαράδεκτο όπως θεωρώ εγώ. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής έχετε τον λόγο. Αληθεύει κύριε Σούλτ ότι η συνθήκη της Λισαβόνας δεν επιτρέπει την χρηματοοικονομική ανάληψη χρεών από τα κράτη-μέλη άλλων κρατών ανάληψη χρεών και έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται πλήρως ευθυγραμμισμένη με την συνθήκη σέβεται απόλυτα το πλαίσιο της συνθήκης γνωρίζω τη συζήτηση που διεξάγεται στη Γερμανία και σε άλλα κράτη-μέλη και θα ήθελα να πω ότι είναι λάθος, απλά λάθος αυτό το οποίο ε, να εξετάζουμε να χαρακτηρίζεται ως bailout δεν είναι bailout. Είναι συνδυασμός δυνατοτήτων ε, και από πλευράς ε, νομικών ευκαιριών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβλέπει, επιτηρεί τα πράγματα. Πρέπει με δημιουργικό, με φάνταστο τρόπο μετά από τις εκτενείς συζητήσεις με τα κράτη-μέλη να μπορέσουμε να δράσουμε. Απόλυτα ευθυγραμμίζεται όμως με τις συνθήκες και απόλυτα με τους όρους του παιχνιδιού. Και κατά τα άλλα το βρήκα αξιοπρόσεκτο ήταν τόσο δύσκολο να βρεθεί μια λύση με αλληλέγγυο τρόπο προς την Ελλάδα όταν, όταν μπορούσε να εξευρεθεί για την ε, Λετωνία, την ε, Ουγγαρία, τη Ρουμανία. Αν δεν μπορούμε να βρούμε μια λύση αλληλεγγύης ε, και ε, βοήθειας, τότε θα πρέπει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να δώσουμε αυτή τη βοήθεια εκτός Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης, τότε στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Καταλαβαίνω ότι προσπαθείτε να παρακάμψετε την απάντηση στην ερώτησή μου γιατί είναι δυσάρεστη η ερώτησή μου. Την επαναλαμβάνω Επαναλαμβάνω λοιπόν, υπάρχει τουλάχιστον η δυνατότητα κράτη-μέλη όταν τα ίδια <clears throat> μπορούν να λαμβάνουν χρήματα για βελτιωμένους, ε, ε, με βελτιωμένους όρους κάποιες χώρες που δίνουν χρήματα να έχουν κέρδος. Αν λέει η ρήτρα bailout clause ότι δεν μπορεί κανείς να αναλάβει τα χρέη ενός άλλου κράτους δεν επιτρέπει να υπάρχει ε, κέρδος από την παροχή χρημάτων σε ένα κράτος. Είσαστε πρόθυμος να συζητήσετε αυτό το θέμα με τον κύριο Σαρκοζή, με την κυρία Μέρκελ, αυτή την υπόθεση παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής έχετε τον λόγο. Συζητούσα αυτό το θέμα επί πολλέ εβδομάδε με του αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων και μπορώ να σα το πω αυτό ειλικρινά κύριε Σούλτ. Και δυστυχώ η μόνη εφικτή λύση ήταν αυτή, αυτή που υιοθετήθηκε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευθύ εξ αρχή ζητούσε να υπάρχουν πιο χειροπιαστά μηνύματα αλληλεγγύη προ την Ελλάδα. Φυσικά πάντα σεβόμενη την αρχή της ε, ε, υπευθυνότητας ε, και του επιμερισμού της ευθύνη Όμως αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μπορέσει να επιστρέψει στην χρηματοοικονομική ομαλότητα η Ελλάδα. Και η λύση που βρέθηκε ήταν αυτή ότι θα δώσουν τα κράτη-μέλη στην Ελλάδα δάνεια από πλευρά τους ε, ε, με ευνοϊκά επιτόκια και όχι υπερβολικά επιτόκια. Και έτσι με τη δημιουργία αυτών των όρων δανεισμού θα μπορέσουν τα πράγματα να λειτουργήσουν για να βοηθηθεί η Ελλάδα. Ευχαριστώ. Πολύ σας ευχαριστώ. Γκίφα Χόφστατ, εξ ονόματος των Φιλελευθέρων Δημοκρατών. Όσον αφορά τη ρήτρα για τη διάσωση, δεν λέει αυτό η συνθήκη. Η συνθήκη λέει ότι δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε να αναλάβει ένα κράτος χρέη άλλου κράτους, αλλά δεν λέει ότι απαγορεύεται κάτι τέτοιο. Αυτό πρέπει να είναι σαφές, γιατί διαφορετικά είναι καταστροφική η ερμηνεία της ε, συνθήκης. Ε, το γράμμα της συνθήκης λέει ότι δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε ένα κράτος μέλος να αναλάβει χρέος. Οπότε, ότι όταν μιλάμε για την Ελλάδα, επί τη βάση της συνθήκης, μιλάμε για πράγματα που είναι δυνατά όταν εφαρμόζεται σωστά η συνθήκη. Τώρα, το 7,6% που είναι πολύ ψηλότερο από το γερμανικό επιτόκιο. Υπάρχουν δηλαδή και άλλα μέτρα που πρέπει να ε, ληφθούν. Πρέπει να υπάρξει μια συγκεκριμένη στρατηγική για τις χρηματοοικονομικές αγορές της Ευρώπης και πολλές μεταρρυθμίσεις. Πότε έχετε σκοπό να παρουσιάσετε ένα πακέτο τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεων δεδομένου από τη στιγμή που υπάρχει το πρόβλημα. Οπότε μπορείτε να μας πείτε πότε θα τεθεί στο τραπέζι του Συμβουλίου ένα τέτοιο είδους πακέτο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φερχόφστατ. Απάντησα και στον κύριο Σούλτς ε, αν υπάρχουν ερωτήματα που θέλετε να θέσετε στην κυρία Μέρκελ, να τα θέσετε στην κυρία Μέρκελ. Εγώ δεν είμαι εδώ για να απαντήσω εξ ονόματος κυρίας Μέρκελ, είμαι εδώ για να απαντήσω εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό το λέω για να είναι σαφή τα πράγματα. Από πλευρά λοιπόν Επιτροπής, Ας είμαστε σαφείς. Η λύση που βρήκαμε ε, σέβεται την ρήτρα της μη διάσωσης, αυτή που ονομάζουμε ρήτρα μη διάσωση. Αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τα μέτρα, η ανακοίνωση και η πρόταση που θα κάνουμε ε, αναμένονται τον επόμενο μήνα. Θα έχουμε την ανακοίνωση για την ε, διακυβέρνηση της Ευρωζώνης, την ισχυμένη διακυβέρνηση και έλαβε όλη η ΡΕΝ εντολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να γίνει συζήτηση με τους Υπουργούς Οικονομικών. Πιστεύω λοιπόν ότι κατά, το διάρκεια, κατά τη διάρκεια του μηνός Μαΐου θα γνωρίζετε ε, την ουσία των προτάσεών μας για την ενίσχυση της ε, διακυβέρνησης στο πλαίσιο της Ευρωζώνης. Ευχαριστώ συμπληρωματική ερώτηση, κύριε Σφερχόφσταντ. Ε, το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, αυτή η ιδέα ε, του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου θα είναι τμήμα τη πρόταση αυτή. Ε, μία απόφαση πολύ συγκεκριμένη γι' αυτό ε, μπορώ να σας πω το εξής, ότι ο στόχος μας είναι να μην ε, ιδρύσουμε ένα νέο ακόμη οργανισμό ε, στο πλαίσιο της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης. Μπορώ να σας πω ότι μπορούμε να σκεφτούμε την ιδέα μιας διευκόλυνσης. Κάτι τέτοιο μου φαίνεται με ένα καλή ιδέα και προσπαθούμε τώρα να διερευνήσουμε τις ε, διάφορες ιδέες ε, που υπάρχουν για να ενισχύσουμε και να ιδρύσουμε ενδεχομένως νέους μηχανισμούς ε, εγγυήσεων όπως αυτούς που θα, προ, που θα πρόβλεπε ο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Κύριος Κομπεντήτ. εγώ θα ήθελα να μας πει ε, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να ε, δανείσει στο επιτόκιο που θα έπρεπε να δανείσει. 3% αλλά δεν μπορείτε να μας το πείτε αυτό βεβαίως. Όσον αφορά τώρα την άκτα, από το 2008 διαπραγματεύεστε το θέμα αυτό της παραχάραξης και της πειρατείας. Υπήρξε ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Μάρτιο προς την κατεύθυνση της μείωσης των διαπραγματεύσεων για το θέμα ακριβώς της ε, παραχάραξης. Ένα χρόνο το περιμένουμε αυτό. Ένα χρόνο. Ε, την αξιολόγηση των συζητήσεων και ένα κείμενο μετά από την Σύνοδο της Νέας Ζηλανδίας. Αυτό που σας ζητώ και το γνωρίζετε είναι... Ε, να ξέρετε ότι εμείς θα πρέπει να πούμε ναι ή όχι στο τέλος των διαπραγματεύσεων. Εμείς δεν θα πρέπει να συμμετέχουμε εμείς καλύτερα από την αρχή για να είναι και πιο διαφανείς οι διαπραγματεύσεις. Γιατί διαφορετικά θα βρεθείτε με το κοινοβούλιο αυτό στην ίδια κατάσταση ε, που βρεθήκατε και με το SWIFT. Σας ζητώ λοιπόν από τώρα κιόλα περισσότερη διαφάνεια να μας δώσετε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε από τώρα ε, όπως γίνεται και με τις, ε, στο των μεγάλων επιχειρήσεων διαχειρίζουν όταν γίνονται διαπραγματεύσεις. Κοιτάξτε, έχω το μεγαλύτερο σεβασμό για το Κοινοβούλιο, κύριε Κομπεντίτ. Γι' αυτό ακριβώς ε, ο Κάρελ Ντεγκούχ, το Επίτροπος, ε, ζήτησε να μπορούν να είναι δημόσια όλα τα κείμενα των διαπραγματεύσεων για να δημοσιοποιηθούν όπως το γνωρίζετε και εσείς στις 21 Απριλίου. Αυτές οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν πριν από την έναρξη ισχύω της συνθήκης της Λισαβόνας και αυτό το γνωρίζετε βεβαίως και επίσης ε, έχουμε ιδιαίτερο συμφέρον να συμμετέχει και το Κοινοβούλιο δεδομένων των νέων, συνθηκο... των νέων εξουσιών που έχει το Κοινοβούλιο και εμείς είμαστε υπέρ ε, μιας αύξησης συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, σε ζητήματα που αφορούν και διεθνείς υποθέσεις. Κοιτάξτε, δεν πρέπει να παίζουμε με τις λέξει, λέει ο κύριο Κομπεντίτ. Αν δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν μπορούν να συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις, δεδομένου ότι υπάρχει συνθήκη της Λισαβόνας πλέον. Δεν είναι ζήτημα λοιπόν να ζητήσετε απλώ από του εταίρου σα να δημοσιεύσουν τα πρακτικά για το κοινοβούλιο. Πρέπει να το κάνετε, υποχρεούστε να το κάνετε, γιατί διαφορετικά το κοινοβούλιο δεν θα πει ποτέ ναι, γιατί έχουμε περάσει συνθήκη τη Λισαβόνα. Είστε υποχρεωμένο λοιπόν να έχετε διαφάνεια ε, στι σχέσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διαφορετικά, ε, αν θεωρείτε ότι θα είναι ναι η απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να μην είστε και πολύ σίγουρο. για την έναρξη ισχύω συνθήκη τη Λισαβόνα. Κοιτάξτε, εγώ υποστηρίζω την ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου Έπρεπε να ζητήσουμε όμω έπρεπε να πάρουμε την άδεια των εταίρων, ε, των, ε, των εταίρων μας τη διαπραγματεύσεις. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν ορισμένε διεθνεί διαπραγματεύσει, οι οποίε είναι κάπω πιο ευαίσθητε και πρέπει για συγκεκριμένου τομεί ε, να έχουμε κάποιε επιφυλάξει. Αλλά προσπαθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο να εμπλέξουμε το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο τη συνθήκη τη Λισαβόνα και σε αυτά που, στο πλαίσιο αυτών προβλέπει για τι διεθνεί διαπραγματεύσει. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρου των ε, συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Κύριε Πρόεδρε, εν ώψη της αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, ε οδηγία για του εργαζομένου, αποφασίστηκε να διαγραφεί η ρήτρα opt-out από την οδηγία. Όπως θα θυμάστε, οι ευρωβουλευτές ε, των εργατικών ζήτησαν να διαγραφεί η ρήτρα opt-out παρά το γεγονό ότι η κυβέρνησή του δεν είχε ζητήσει κάτι αντίστοιχο. Τώρα έχουμε μια περαιτέρω αναθεώρηση και οι Ευρωπαίοι θέλουν οι πολίτε του να μπορούν να εργάζονται σε πιο ευέλικτα ωράρια. Και φαντάζομαι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει κάτι το οποίο θα σέβεται τα ευέλικτα ωράρια τη εβδομάδα ε, των 48 ώρων. Δεν έχω ακόμα ένα σχέδιο οδηγία ε, νομοθετική πρόταση δεν έχω καμία ιδέα για την ουσία των αλλαγών. Όπως ξέρετε υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο είναι ανοιχτό σκοπίμως. Θέλω να ακούσω και τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων, διότι οι νέοι κανόνες θα πρέπει να προστατεύουν τους εργαζομένους από υπερβολικά ωράρια εργασίας και θα πρέπει να τους δίνεται και χρόνος ανάπαυσης. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει συμφωνία μεταξύ οικογενειακής και εργασιακής ζωής και κυρίως να λαμβάνουμε υπόψη και τα ωράρια των εργαζομένων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιε μέρημνε, διότι ξέρετε ότι υπάρχουν ε, και αποφάσει δικαστηρίων που μα υποχρεώνουν να βρούμε μια λύση. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν κάτι για τη νέα λύση και θα ε, αποφύγουμε τη μακροσκελή συζήτηση που δεν μα επέτρεψε να καταλήξουμε σε λύση την προηγούμενη φορά. Κατανοώ ότι ο πρόεδρο ε, Μπαρόζο δεν θέλει να προκαταβάλει το αποτέλεσμα τη οδηγία, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 3 εκατομμύρια άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο που ε, απολαμβάνουν αυτή τις ρητρες opt opt-out και πραγματικά ε, δεν ξέρουν τι να πούνε στο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να δυσκολέψει τη ζωή τους. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά φαντάζομαι ότι θα προσπαθήσετε να κάνετε κάτι αυτή τη φορά για να λύσετε το θέμα. Είστε πολύ ευγενικό κύριε Κύρκο, αλλά πέραν της ε, Βρετανίας υπάρχουν και άλλα 26 κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατανοείτε λοιπόν ότι παρά το γεγονό ότι κατανοούμε πάρα πολύ καλά το θέμα τη συνένεση που έχετε πει, αλλά θα πρέπει να ακούσω και άλλε νομοθετικέ ανησυχίε. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα και θα πρέπει να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ τη ευελιξία, την οποία εσεί επισημαίνετε για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, αλλά και τη προστασία των εργαζομένων. Και αυτό θέλουμε να το κάνουμε. Αυτό ε, θέλουμε να κάνουμε, γι' αυτό κάνουμε και έκκληση και στους κοινωνικούς εταίρους για να έχουμε μια επικοδομητική πρόταση. Ο κύριος Μπίσκι, εξ ονόματος της Ενωμένης Αριστεράς. ευχαριστώ κύριε ε, Ευχαριστώ κύριε Μπαρόζο. Μιλήσατε για το πρόγραμμα εργασιών που συζητήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είπατε ότι κριτικές παρατηρήσεις θέλετε να τύχουν συνέχεια και να εξεταστούν. Έχω μία ερώτηση όμως. Έχει γίνει πολλής λόγος για την κρίση και το ξεπέρασμα της κρίσης και την αντιμετώπιση της. Έχω όμως την εντύπωση ότι όσα έγιναν σε σχέση με τις τράπεζες λίγα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Μία ερώτηση θα με ενδιέφερε. Νομίζετε ότι κάνατε επαρκή πράγματα, έκανε επαρκώς το, η δουλειά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τι χρειάζεται να γίνει θα λέγατε ώστε τα αίτια τη ε, χρηματοοικονομική κρίση να καταπολεμηθούν ώστε η πρακτική των τραπεζών να μην τύχει συνέχεια όπω έγινε μέχρι σήμερα. Um, Σα ευχαριστώ. Σήμερα κιόλα μόλις ε, υποβάλαμε στο πρόγραμμα εργασιών μας την δράση μας ε, για τον χρηματοοικονομικό τομέα. Έχουμε κάνει ένα σημαντικό μέρος της δουλειάς, απομένει να γίνει ακόμα ένα άλλο σημαντικό μέρο της δουλειάς. Είναι σωστή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λέγω και λυπούμε ότι μειώθηκε το επίπεδο φιλοδοξιών από τα κράτη-μέλη όσον αφορά ένα πλαίσιο ε, εποπτείας το οποίο εξετάζετε τώρα εσείς ως πρόταση και θα έχουμε σε σχέση με τις προτάσεις που θα υποβληθούν στο Κοινοβούλιο ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε. Υπάρχουν όμως κάποια πιο συγκεκριμένα θέματα που μπορούν να γίνουν, πιο χειροπιαστά. Υποστηρίζω για παράδειγμα ένα τέλος που θα πρέπει να εισπράτεται από τις τράπεζες. Είναι θέμα για τη λέσχη των 20, την G20. Είναι δίκαιο και σωστό ο τραπεζικός τομέας μετά από όλα τα προβλήματα που δημιούργησε να συνεισφέρει και αυτός από πλευράς του για να επιληθούν τα προβλήματα σε σχέση με το μέλλον των οικονομιών μας. Είναι θέμα ισορροπιών. Δεν θέλουμε να υπονομεύσουμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, τον τομέα τον τραπεζικό δηλαδή, όμως πιστεύουμε ότι περαιτέρω μέτρα είναι αναγκαία και είναι σημαντικά για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο χρηματοοικονομικό τομέα. Κύριε Μπαρόζο, μια σύντομη επερώτηση έχω ο κύριος Σάκερμαν ε, δύσκολα εντυπωσιάζεται. Έκανε λόγο απλά 25% κέρδους ε, να μπορούν να πετύχουν οι τράπεζες. Δεν είναι αυτό υπερβολικά υψηλό σύμφωνα με την άποψή σας ε, δεδομένων των μέτρων. Δεν αλλάζει τίποτα. Θέλει πάλι 25% μερίσματα όσον αφορά το κέρδος. Ο κύριος Σάκερμαν, ο πρόεδρος της Γερμανικής Τράπεζας, δεν είναι κάποιος ασήμαντος αυτός και οι απόψεις του. Σας ευχαριστώ. Λυπούμε, δεν παρακολούθησα τις δηλώσεις του Προέδρου της Deutsche Bank, της ε, Γερμανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να σχολιάσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Η Ευρώπη της ειρήνης και της δημοκρατίας. Ο κύριος από Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λόγω αυτής της κρίσης ε, που ήταν τραπεζική και πιστοτική και που απέρευσε από τις μεγάλες εμπορικές ε, ε, τράπεζες στην Σκοτία για παράδειγμα, δέχεστε ότι εναλλακτική σε δυνατότητες για την διαχείριση αυτών των αποταμιεύσεων είναι κάτι το οποίο έχει λάθος στόχους και είναι μια πρωτοβουλία η οποία δεν είναι θετική από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και που στοχεύει στον απόλυτα λάθος στόχο. Καθόλου, λέει ο κύριος Μπαρόζο. Είναι μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία. Ακριβώς επειδή ο στόχος είναι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη σε ένα πάρα πολύ σημαντικό τομέα των οικονομικών αγορών μας. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον του οικονομικού τομέα να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη. Ας το δούμε αυτό. Υπάρχει πρόβλημα εμπιστοσύνης, αξιοπιστίας στο χρηματοοικονομικό τομέα. Αυτό έχει τις ρίζες του στην ανεύθυνη στάση κάποιων μεγάλων τραπεζών και σε άλλες χώρες, ε, στη είπα και αλλού και μεγάλο μέρος αυτής της κατάστασης ε, είχε τις ρίζες του στις ΗΠΑ. Πρέπει να βρεθούν σωστές ρυθμίσεις. Πιστεύουμε ότι οι ρυθμίσεις που προτείνουμε αποκαθιστούν ε, τη σωστή ισορροπία και δεν στοχεύουν στο να δημιουργήσουν δυσκολίες στον χρηματοοικονομικό τομέα καθόλου. Το αντίθετο θέλουν να διευκολύνουν διότι χρειάζεται αυτή την αξιοπιστία ο χρηματοοικονομικός τομέας για να χρηματοδοτήσει την οικονομία. Πρόεδρε, επερώτηση. Πώς η οδηγία του AIFM μπορεί τους διαχειριστές των εναλλακτικών ταμείων να συνεισφέρει για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης όταν το πρόβλημα είναι σε σχέση με τις εμπορικές τράπεζες. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Πρόεδρος Μαρόζο. δεν, λυπούμε αλλά δεν συμφωνώ ότι το πρόβλημα είναι μόνο των τραπεζών. Πράγματι τα προβλήματα στις ΗΠΑ δεν δημιουργήθηκαν μόνο από τις μεγάλες τράπεζες, προκλήθηκαν επίσης και από μη εμπορικέ τράπεζες, από ενώσεις επενδυτικές και hedge funds. Δεν συμφωνούμε με την ανάλυση σας ότι οφείλονται όλα αυτά μόνο στις μεγάλες εμπορικές τράπεζες. Μάλιστα κάποιες από αυτές δεν ήταν ακριβώς υπεύθυνε για αυτήν την κρίση. Οι εμπλεκόμενοι στην αγορά έχουν συγκεκριμένες ευθύνες. Δημιουργήθηκαν προβλήματα στον χρηματοοικονομικό νομικό τομέα. Και ο τομέας ε, των νομικών ρυθμίσεων είναι το πιο εύθετο πεδίο δράσης για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τα πράγματα και την εμπιστοσύνη του στις αγορέ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Ο Άντριο Χενρί Μπρόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε η Ευρωπαϊκή Διπλωματική Υπηρεσία θα, είναι, θα λογοδοτεί στον ανώτατο εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική. Ο ρόλος σύμφωνα με το άρθρο 18 του ανώτου είπα του εκπροσώπου είναι να καθορίζει την εξωτερική πολιτική όπως σύμφωνα με τις εντολές του Συμβουλίου. Και φυσικά στο Συμβούλιο υπάρχουν εκπρόσωποι των κρατών μελών. Όμως υπάρχουν σχόλια μεταξύ των πολιτικών ομάδων που θέλουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην διπλωματική υπηρεσία. Ιδιαίτερα λέγοντα ότι 50% θα πρέπει των υπαλλήλων τη εξωτερική αυτή διπλωματική υπηρεσία να καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και δεν θα πρέπει από διακυβερνητικό πλαίσιο ε, intergovernmentalism, ζητώ συγγνώμη για τη χρήση αυτού του όρου, αλλά αφορά το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτό. Επιπλέον, είπατε εκπρόσωπο, ε, όντα αντιπρόεδρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πω αυτό δείχνει ότι πρέπει να κινηθούμε. Αυτό δείχνει ότι η εξωτερική πολιτική θα πρέπει να ε, είναι στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι πραγματικά μύθος ότι η ύπατος εκπρόσωπος ε, ε, ακολουθεί την εξωτερική πολιτική με εντολή του Συμβουλίου. Συμφωνείτε με αυτό. Όχι πράγματι η δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου και του αξιώματος του είπα του εκπροσώπου είναι μία από, ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της συνθήκης Λισαβόνας. Και αυτό που θέλουμε είναι σε σχέση με τις κυβερνητικές αρμοδιότητες και τις κοινοτικές αρμοδιότητες να υπάρξει η σωστή ισορροπία. Η ΚΕΠΑ θα είναι ουσιαστικά διακυβερνητικού χαρακτήρα. Αυτό είναι δικαίωμα, είναι προνόμιο των κρατών μελών. Υπάρχουν όμως άλλα κινητικά θέματα τα οποία δεν θα πρέπει να εντάσσονται στο διακυβερνητικό πλαίσιο. Θα πρέπει να παραμένουν σε κοινοτικό επίπεδο πάντως εκπρόσωπος λοιπόν αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, έχει διτή ιδιότητα. Θα πρέπει με αυτές τις ε, αρμοδιότητες που έχει υποσυνέργεια να χρησιμοποιεί και τα δύο σκέλη των αρμοδιοτήτων της. Θα υπάρχουν αρμοδιότητες φυσικά που θα μπορεί να αναπτύξει εντό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω αντιπρόεδρο τη Επιτροπή, αλλά θα μπορεί να συνεργάζεται και να ευθυγραμμίζεται με τα κράτη-μέλη στη συνεργασία αυτή μέσα στο πλαίσιο των εντολών του Συμβουλίου. Αυτό είναι ο στόχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ενισχύσουμε την προάσπιση των συμφερόντων μα και να προαγάγουμε τι αξίε μα παγκόσμια. Σα ευχαριστώ. Επερώτηση κατανοώ την συνεκτικότητα την εσωτερική, στο εσωτερικό πλαίσιο λόγω της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που στοχεύεται να επιτύχετε. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε την συνθήκη της Αβώνας που είναι αρκετά αρνητική και σχεδόν να αποκλειστεί το Συμβούλιο που τουλάχιστον παρόλα τα ασφάλματα έχει εκπροσώπους των κρατών μελών το Συμβούλιο δεν θα μπορούσα ποτέ να πω ότι θα πρέπει να παραβούμε τις συνθήκες, διότι καθήκον μας είναι να είναι σεβαστή η συνθήκη, οι συνθήκες και οι διατάξεις. Αυτό ζητούμε λοιπόν, να είναι σεβαστή η συνθήκη και η συνθήκη καθορίζει μια ισορροπία. Και αυτή η ισορροπία πρέπει να είναι σεβαστή. Είναι μια πρόοδος σε σχέση με το παρελθόν αυτό, όπου τελείως διαφορετικά <clears throat> θεσμικά όργανα <clears throat> καλούνται να δημιουργήσουν ένα κοινό πλαίσιο προ τα κοινά συμφέροντα υπέρ των ευρωπαϊκών αξιών παγκόσμια. Είναι δυνατόν, σεβόμενοι τι συνθήκε, να πετύχουμε αυτό το οποίο ακριβώ θέλει να πετύχει η συνθήκη. Και αυτό μπορεί να γίνει σε ένα πνεύμα καλή συνεργασία μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων και με σεβασμό φυσικά και των πολιτικών των κρατών μελών και των στόχων του. Σας ευχαριστώ, λέγει ο Πρόεδρο. Ολοκληρώσαμε τώρα τον γύρο των ε, γενικών ερωτήσεων. Ας περάσουμε τώρα σε πιο εξειδικευμένο θέμα. Την κατάσταση όσον αφορά την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Σιλβέστρης θα είναι ο πρώτος που θα πάρει. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Εγώ κατάγομαι από τον Νότο στην Ιταλία και η δική μας οικονομία βασίζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην κλωστοϊφαντουργία, στην υποδηματοπία και σε τέτοιου τύπου επιχειρήσεις και στη γεωργία φυσικά. Δυστυχώς οι κλάδοι αυτοί αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα από τις αγορές που προέρχονται από την Κίνα και τις υπόλοιπες αναστατικές χώρες. Ένα υπόδημα μπορεί να στοιχίζει 30 ευρώ ε, στην Ιταλία και όταν προέρχεται από την Κίνα στοιχίζει 10 ευρώ. Ένα μικρό μπουκαλάκι για παιδάκι στοιχίζει 4 ευρώ σε εμά και όταν έρχεται από την Κίνα στοιχίζει 1 ευρώ. Όταν λοιπόν συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα, χάνονται χιλιάδε θέσει εργασία και υπάρχει φυσικά και εγκατάλειψη τη περιοχή. Όταν ε, ε, συναντώ λοιπόν ε, μικρού ε, βιοτέχνε, μου λένε τι περιμένετε, γιατί δεν τα φορολογείτε, γιατί δεν τα σμαλογείτε όλα αυτά. Τα παιδιά στην Κίνα δουλεύουν ε, από μικρή ηλικία χωρί καμία ασφάλεια, χωρί καμία πρόνοια και καμία προστασία. Ποια είναι η λύση. Όταν εγώ συναντώ του επιχειρηματίε, τι μπορώ να του πω ότι κάνει η Ευρώπη για μια κρίση η οποία είναι μη αναστρέψιμα. Χάνουμε τεράστιο αριθμό θέσεων εργασία, όλα γίνονται καπνό και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πώ μπορούμε να σώσουμε την Νότια Ιταλία, διότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Χρειάζομαι απαντήσει, κύριε Επίτροπε, και τι θέλω από εσά. Ευχαριστώ. Κατανοώ τι ανησυχίε σας, ε, καθόλου λογικέ. Και θα ήθελα να πω κάποια πράγματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι όπως ξέρετε είναι ο κινητήριος μοχλός για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Πώ μπορούμε να απαντήσουμε λοιπόν στο θέμα του ανταγωνισμού που προέρχεται από άλλε περιοχέ εκτό Ευρωπαϊκή Ενώσεω που έχουν πολύ χαμηλέ προδιαγραφέ ε, και για την ε, προστασία των εργαζομένων και για το περιβάλλον. Η λύση δεν είναι να κλείσουμε τα σύνορά μα σε καμία περίπτωση γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερο εξαγωγέα ανά τον κόσμο. Η λύση είναι να προάγουμε την αξιοπρεπή εργασία και να υπάρχουν συγκεκριμένα πρότυπα και προδιαγραφέ ανά τον κόσμο. Αυτό προσπαθούμε να το πιέσουμε στο G20, στη Διεθνή Οργάνωση εργασία. και αυτό είναι και τμήμα του διαλόγου που έχουμε με τους εταίρους μας. Και δεν θεωρώ βέβαια ότι θα μπορούσε να υπάρξει λύση εάν δεν χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένα μέτρα αντι-dumping. Δεν είναι λύση το να κλείσουμε τα σύνορά μας ε, ενώπιον πολύ σημαντικών εμπορικών εταίρων. Θα είναι καταστρεπτικό για μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιώργος παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, με αφορμή την διαχείριση του ελληνικού προβλήματο έγιναν και προηγουμένω αναφορέ, Για όλου εμά που παρακολουθούμε από κοντά την εξέλιξη ε, και τη διαχείριση του προβλήματο, αντιλαμβανόμαστε και έχουμε μια αίσθηση αρκετοί από εμά παραγωνισμού τη Επιτροπή από το συμβούλιο. η επιτροπή ήταν ανέκαθεν νομίζω εξορροπητικό παράγοντα των μεσαίων και μικρότερων κρατών μελών της ένωσης έναντι του συμβουλίου και σήμερα νομίζω ότι ο ρόλος της στα θέματα που ε, αντιμετωπίζει η ελλάδα και όχι μόνο περιορίζεται σε τεχνοκρατικές κινήσεις και δηλώσεις. ρωτάω λοιπόν συγκεκριμένα μιλάμε για την οικονομία μιλάμε για την νομισματική ένωση όπου τα υπερεθνικά στοιχεία θα είναι εντονότερα και εν ώψη και της φιλόδοξης στρατηγικής ε, για το 2020 που καταρτίζει η επιτροπή αναφερόμαστε στην καταπολέμηση της ανεργίας στην καταπολέμηση της φτώχειας πώς όταν η επιτροπή δεν έχει το ρόλο που της αρμόζει θα μπορέσει να υλοποιήσει αυτές τις φιλόδοξες στρατηγικές. Το ζήτημα της απασχόλησης ε, γνωρίζετε ότι εξαρτάται από την ευρύτερη οικονομική κατάσταση. Πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς γι' αυτό. Δεν μπορούμε να αποκαταστήσουμε τα επίπεδα απασχόλησης που είχαμε πριν από την κρίση, πριν ε, να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε ρυθμούς ανάπτυξης. Γι' αυτό ακριβώς ε, χρειαζόμαστε νέες πηγές ανάπτυξης και προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε ε, τους τομείς που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι μία προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή. Όπως είπατε κι εσείς, ε, έχουμε συγκεκριμένα προγράμματα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ε, Στρατηγικής για το 2020, ε, νέα προγράμματα για τους νέους, αλλά η βασική μας προτεραιότητα είναι να αποκαταστήσουμε τις συνθήκες, την εμπιστοσύνη στην οικονομία και γνωρίζετε κι εσείς λόγω του προβλήματος στην Ελλάδα ότι το θέμα της εμπιστοσύνη στην οικονομία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρώτα πρέπει να, να καλύψουμε τις ε, δημοσιονομικές ανισορροπίες. Ο κύριος Δορντών. No. Frederic Dordon, please. Monsieur le Président, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση της απασχόλησης είναι πολύ, πολύ ανησυχητική. Το 2009 2,7 ε, εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη δουλειά τους. Ε, αυξάνεται σε 8% ο μέσος όρος της ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και περίπου 17% ε, του πληθυσμού ζει στο κατόφλι της φτώχειας. Μήπως νομίζετε λοιπόν ότι μια στρατηγική που θα βασίζεται σε δύο βασικούς άξονες πρέπει να υπάρξει πρώτον ενίσχυση της αξιοπρεπούς εργασίας ε, και η στρατηγική 2020 μήπως θα έπρεπε να ασχολείται με αυτήν τη θεματική ενότητα και όχι τόσο με την ανάπτυξη όσον αφορά την ε, αηφόρο και αλληλέγγυη ανάπτυξη. Πώς έχετε σκοπό να ενισχύσετε την ε, πράσινη απασχόληση και την ευφύη απασχόληση δίνοντας ιδιαίτερη σημασία κυρίω ε, στην απασχόληση των νέων, το αναφέρατε αυτό, αλλά και όσων έχουν, ε, είναι πάνω από 50 ετών. Η αύξηση της ε, ζήτησης, η παγκοσμιοποίηση ζητούν νέε πολιτικές στο πλαίσιο το παγκόσμιο. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, τα προβλήματα αυτά έχουν συμπεριληφθεί στη στρατηγική για το 2020. Είχα αναφέρει το θέμα αυτό στο πλαίσιο των πολιτικών κατευθυντηρίων γραμμών, αλλά είναι πολύ σημαντικό και το ζήτημα της νέας, της πολιτικής, της βιομηχανικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχουμε μια ε, βιο, ε, βιώσιμη, πιο εξυγχρονισμένη βιομηχανική πολιτική. Ε, επίσης, έχουμε για τους νέους πολλές πρωτοβουλίες, όπως ε, για παράδειγμα αυτή που αφορά τις νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας και θέσαμε ε, δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή σε ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση, την ε, καταπολέμηση της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα σημεία όλα στην στρατηγική για το 2020, ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι η καταπολέμηση της ανεργίας είναι πρώτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι η ανάπτυξη της στρατηγικής αυτής θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε σημαντικά αποτελέσματα για την καταπολέμηση της ανεργίας. Ευχαριστώ πολύ. Ο Σέντζιο Κοφεράτη. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε, η ανεργία αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, και λόγω στοιχείων που διαφέρουν το ένα από το άλλο και κατά πάσα πιθανότητα θα αυξηθεί στα επόμενα χρόνια κι άλλο. Πολλοί εμπειρογνώμονε λένε ότι θα χρειαστούμε τουλάχιστον δύο χρόνια προκειμένου τα, οι ενδείξει ανάκαμψης που αρχίσαμε να διαπιστώνουμε να γίνουν ε, πραγματικότητα και ότι για τα επόμενα δέκα χρόνια η ανάκαμψη θα είναι τόσο αργή που δεν θα δημιουργηθούν επιπλέον θέσεις εργασία. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε αύξηση τη ανεργία, θα χάνει τη θέση εργασία του όποιο αυτή τη στιγμή ε, είναι ενεργό ε, πληθυσμό, εργαζόμενο, και οι νέοι που θέλουν να ενταχθούν στην αγορά εργασία. δεν θα μπορούν βρω μια θέση απασχόλησης. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο λοιπόν δεν θα πρέπει να προαχθεί μια δράση για την προστασία του εισοδήματος όλων όσων χάνουν τη θέση εργασίας τους ανά την Ευρώπη και να θεωρήσουμε και τους νέους ως ένα κατεπήγον θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Να έχουμε και στοιχεία κατάρτισης τα οποία ε, θα τους επιτρέπουν ε, να έχουν και τη δυνατότητα να ξαναβρούν μια θέση εργασίας. Έχετε δίκιο στην ανάλυση που κάνετε για την αγορά εργασίας. Πράγματι, η κατάσταση συνεχώς επιδεινώνεται. Παρά το γεγονός ότι είναι λίγο πιο ε, σταδιακά τα βήματα από ό,τι στο παρελθόν, βλέπουμε κάποια στοιχεία ανάκαμψη στα κράτη-μέλη, αλλά έχουν περάσει εννέα μήνες από τότε που άρχισε να ανακάμπτει η οικονομία από την βαθιά ύφεση και θα περάσει και κάποιο χρονικό διάστημα εντός του τρέχοντος έτους, όταν οι ευάλωτοι ε, οικονομική δραστηριότητα αρχίσει να δείχνει σημεία ανάκαμψη. Γι' αυτό λοιπόν και η πρώτη προτεραιότητά μα είναι η ανεργία και κυρίω η ανεργία των νέων όπω είπατε κι εσεί. Έχουμε άνω του 20% των νέων ανθρώπων αυτή τη στιγμή ανέργου ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και ακριβώ ε, ξεκινήσαμε τρει πρωτοβουλίε για το θέμα αυτό. Δύο από αυτέ τι έχω ήδη αναφέρει. Υπάρχει και μια πρωτοβουλία για την ανεργία των νέων και τις θέσεις απασχόλησης για τους νέους και οι πρωτοβουλίες αυτές θα είναι επίσης και μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων κατάρτισης ε, για την επαγγελματική κατάρτιση και υψηλότερε δυνατότητε εκπαίδευση στον χώρο εργασίας μετά από τα, το πτυχίο, τι λεγόμενε εκπαιδευτικέ ε, και ε, περιόδους άσκησης. Ο κύριος Βότσον. Κύριε Πρόεδρε, την περασμένη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κλίματος ξεκίνησε ένα οδικό χάρτη και ένα πρόγραμμα για το 2050. Το πρόγραμμα αυτό δείχνει τρεις τρόπους με τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να μειώσει ε, κατά 20% τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα μέχρι το 2020 όπως ακριβώς ε, ελπίζουμε. Θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα ώστε να είμαστε πλήρως αυτάρκης για τους ενεργειακούς μας πόρους και θα μπορέσουμε να έχουμε και ένα ασφαλές δίκτυο δημιουργίας θέσεων εργασίας και ανάκαμψη της οικονομίας Αυτά όλα βέβαια μπορούν να γίνουν μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εναγκαλίσει αυτό τον οδικό χάρτη, θα κάνει το τόλμημα να προσπαθήσει να δώσει μια νέα όθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία ε, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέτρα και δεδομένου ότι υπάρχουν και δυνατότητε θέσεων εργασία, ε, θα προσπαθήσετε εσεί, ε, κύριε Πρόεδρε να ενθαρρύνετε τα κράτη-μέλη να λάβουν τι ανάλογε δράσει. Τη γνωρίζω την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματο Κλίματος και πράγματι στη στρατηγική για το 2020 έχουμε προτείνει μία ε, πρωτοβουλία για μια αποδοτική Ευρώπη βάσει των πόρων τη, που θα δίνει στην Ευρώπη ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ε, σε σχέση με τους εταίρους της και στόχος αυτός ε, μεταφράστηκε και στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2010 και μετά και προσπαθούμε να έχουμε μία μερική μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλής κατανάλωσης ε, άνθρακα μέχρι το 2050 ε, με συμμετοχή φυσικά και τη μείωση τη κατανάλωση ενέργεια στον τομέα των μεταφορών και κυρίω με επενδύσει. Να τονίσω εδώ τον όρο επενδύσει. Θεωρούμε ότι η πολιτική για το κλίμα όπω δείχνουν και οι ε, δραστηριότητε που έχουμε για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, μία πηγή νέων θέσεων εργασία για του νέου και τι λεγόμενε οικολογικέ εργασίες, πράσινε εργασίε. Η κυρία Χελικά Τρούπελ. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητή Επιτροπή εδώ για νέα μέσα IT όπως ε, ε, τα ηλεκτρονικά βιβλία σε σχέση με την ε, προώθηση προϊόντων σε ψηφιακή μορφή, ιδιαίτερα βιβλίων. Ωστόσο όμως οι περισσότερες αυτές πρωτοβουλίες προέρχονται από τη ΣΥΠΑ. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προαγωγή της ψηφιοποίησης της πολιτισμικής μας κληρονομιάς στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ε, μέσα από την ευρωπαϊκή η δημιουργία των ψηφιακών βιβλίων με την προώθηση ψηφιοποίησης ε, των βιβλίων στις βιβλιοθήκες μας ε, είναι μεγάλη πρόκληση καθιστώντας ε, αυτά τα αγαθά προσπελάσιμα στους ε, πολίτες. Ωστόσο όμως ε, έχουμε και θέματα που αφορούν και εκδότες όσον αφορά τα σπάνια βιβλία Orphan Works. Εδώ θα πρέπει να δούμε σε σχέση με το έργο ότι πρέπει να έρθουμε στο ύψος των περιστάσεων. Εδώ από την Αντιπρόεδρο Κρούς και Επίτροπο Βασιλείου έχει προαναγγελθεί και με χαρά μπορώ να σας το ανακοινώσω ότι ο κύριο Μωρίς Λεβί, η κυρία Ελίζεβεθ Νίγεμαν και ο κύριο Ζακ Ντεκέρκ θα επομιστούν αυτό το έργο. Ω Επιτροπή Σοφών θα προαγάγουν αυτή την ιδέα ώστε η πολύ σημαντική μας πολιτισμική κληρονομιά να προαρθεί σε ψηφιοποίηση σεβόμενη πάντα τα πνευματικά δικαιώματα ε, και τα θέματα προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Μέχρι τα τέλη του έτους θα προχωρήσει. Ο κύριος Σαρνέτσι παρακαλώ, έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ήθελα να μου πείτε τι σύμφωνα με τις απόψεις σας, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις συνολικά στον τομέα των εναερίων μεταφορών λόγω της ε, κατάρρευσης που είδαμε σε σχέση με την ε, διεξαγωγή των ε, αεναέριων μεταφορών η σημερινή εφημερίδα η έκδοση της Financial Times λέει ότι αυτή η κατάρρευση αυτή η κατάσταση που οδήγησε στο να ξεμείνουν χωρίς να μπορούν να ταξιδέψουν πάνω από 7 εκατομμύρια ταξιδιώτες κοστίζει 200 εκατομμύρια δολάρια ημερήσια στους ε, κύκλους των ενέργειων μεταφορών. Ποια θα είναι η επίπτωση στην απασχόληση σε αυτόν τον τομέα. Διότι από ό,τι γνωρίζω αυτό είναι ο πιο σημαντικός ρόλος ε, της ε, απουσίας σας και του κυρίου, της απουσίας του κυρίου Φανρόμπο στην Κρακοβία. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά τον, αυτή την κηδεία στην Κρακοβία θέλω να το διαχωρίσουμε τελείως από τα άλλα θέματα. Έχω πολύ μεγάλο σεβασμό για τον κύριο Κατσίνσκι. Έκανα ό,τι ήταν δυνατό και περνούσε από το χέρι μου για να είμαι παρόν σε εκείνη την κηδεία και όσον αφορά τον θάνατο του κυρίου Κατσίνσκι, της γυναίκας του και όλων εκείνων που ε, σκοτώθηκαν με το αεροπορικό ατύχημα και πραγματικά δεν μπορώ να κατανοήσω πώς είναι δυνατόν να κάνετε τέτοιου είδους επικρίσεις χρησιμοποιώντας ως μέσο το θάνατο τόσων πολλών ατόμων για να ασκήσετε επικρίσεις σε ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο. Το πρόβλημα είναι ότι πολύ αργά το βράδυ μου έδωσαν την πληροφορία ότι η πτήση που είχε διοργανωθεί από τις βελικές αρχές είχε ακυρωθεί και έτσι δεν ήταν δυνατό για μένα να μεταβώ εκεί. Θέλω να το καταστήσω απόλυτα σαφές αυτό. Απόλυτα κατηγορηματικά σαφές ότι έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου. Όχι μόνο να αποτίσω φόρο τιμή εκεί σε αυτούς τους ανθρώπους όντας παρόν εκεί αλλά με κάθε τρόπο να μπορέσω να φτάσω εκεί. Και αυτό θα ήθελα να καταχωρηθεί στα πρακτικά και θα ήθελα σε σχέση με τον τομέα των ε, εναέριων μεταφορών να πω ότι γνωρίζουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ σημαντική επίπτωση αυτή τη έκρηξη αυτού του ηφαιστείου στι εναέριε μεταφορές. Γι' αυτό ήδη προσπαθούμε να θέσουμε εντάξει τα του οίκου ε, να αναλάβουμε δράση για να δούμε τι μπορεί να γίνει, να βοηθήσουμε τι ε, εταιρείε των αερομεταφορών. Σοβαρότατε απώλειε έχουν υποστεί επειδή δεν μπορούν να, κάνουν, να ακολουθήσουν τι εμπορικέ του δραστηριότητε επί πολλέ ημέρε. Πρέπει να βρεθεί μια συνολική σφαιρική λύση για την αντιμετώπιση αυτή τη κρίση. Και πραγματικά αυτή η κρίση μετά την 11η Σεπτεμβρίου είναι η πιο σοβαρή κρίση που αντιμετωπίζουμε. Πρέπει να, δούμε, να βρούμε τρόπου ε, για να ανακουφίσουμε την κατάσταση. Το έχουμε συζητήσει στο ε, Σώμα των Επιτρόπων, ε, στην Επιτροπή, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ο κύριος Νικό, Νικόλαος Χουντής παρακαλώ. Κύριε Μπαρόζο, το 2000 έως το 2006, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση κινήθηκε μεταξύ 8 και 9% προς δόξα της στρατηγικής της Λισαβόνας που μιλούσε για την πλήρη απασχόληση. Πρόσφατη έκθεση της Κομισιόν μιλάει το 2010 ότι η ανεργία θα φτάσει στο 10% και θα το ξεπεράσει ένα κοινωνικό ηφαίστειο για να μιλήσουμε με την ορολογία της περίοδου. Και τρίτο, σε μια σειρά χώρες που εφαρμόζονται προγράμματα λιτότητας όπως στην Ιρλανδία και στην Ελλάδα αλλά και σε χώρες όπως η Ρουμανία, η Ουγγαρία και η Λετωνία που έχει εμπλακεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχουμε αύξηση της ανεργίας σε επίπεδα ρεκόρ. Κατόπιν τούτου, σας ερωτώ, έχει μελετήσει η Κομισιόν τις επιπτώσεις που έχουν αυτές οι πολιτικές λιτότητας τις οποίες και εσείς και οθείτε και πιέζετε χώρες να πάρουν προκειμένου να βγουν από την κρίση έχετε μελετήσει τις επιπτώσεις στην απασχόληση και στην οικονομία μιας χώρας όταν εμπλέκεται το διεθνές νομισματικό ταμείο; πιστεύετε ότι θα μειωθεί η ανεργία στην ευρώπη με αυτές τις πολιτικές; uh, δεν υποχρεώνουμε κανέναν να λάβει μέτρα. Όσον αφορά την Ελλάδα, οι αποφάσει ελήφθησαν από τι ε, Καταλαβαίνετε βέβαια ότι η κατάσταση αυτή των μικροοικονομικών ανισορροπιών στην ελληνική οικονομία είναι πάρα πολύ αρνητική και για την ανάπτυξη αλλά και για την απασχόληση. Είναι σαφές λοιπόν ότι χωρίς να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην, στα δημόσια οικονομικά της Ελλάδος δεν υπάρχει δυνατόν να υπάρχει ανάπτυξη στην Ελλάδα και φυσικά χωρίς την ανάπτυξη δεν μπορούμε να έχουμε νέες θέσεις εργασίας. Δεν θα πρέπει λοιπόν να έχουμε την μακροοικονομική σταθερότητα και να την αντιπαραβάλλουμε με την ανάπτυξη. Το θέμα είναι να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε μια μετάβαση, πώς μπορούμε να έχουμε κίνητρα στην οικονομία και να έχουμε το περιθώριο να γίνουν αυτά και επίσης να σεβαστούμε τι απαραίτητε ισορροπίε τη μακροοικονομική σταθερότητα. Γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο θεωρώ ότι είναι προ το συμφέρον τη ελληνική οικονομία και των Ελλήνων εργαζομένων να έχουν το συντομότερο δυνατό αποκατάσταση αξιοπιστία για τα οικονομικά του. Ευχαριστώ κύριο Πόλη Ρούμπικ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η δική μου ερώτηση αφορά το ηφαίστειο, την έκρηξη του ηφαιστείου, που φυσικά στον τομέα των σωματιδίων σκόνης και στάχτη και των εκπομπών ρήπων διοξιδίου του άνθρακα θα έχει επιπτώσεις. Πιστεύετε ότι είναι δυνατόν να αξιολογηθεί ποια θα είναι η επιβάρυνση μελλοντικά λόγω αυτής της κατάστασης για να μην υπάρξει διακύβευση θέσεων απασχόλησης διότι σε σχέση με την οδηγία κατά των σωματιδίων έχουμε σημαντικού περιορισμού. Ευχαριστώ. Uh, Προσέξτε. Αυτό το πρόβλημα με το ηφαίστειο είναι εκτός ελέγχου σίγουρα είτε από πλευράς ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, είτε από πλευράς ευρωπαϊκών κυβερνήσεων των κρατών μελών. Έχει συμβεί αυτή η έκρηξη και πρέπει να δούμε τώρα τι επιπτώσει. Όσον αφορά τι εταιρείες εναερίων μεταφορών, είπα ήδη ότι εξετάζουμε τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση και με το προηγούμενο το οποίο υπήρχε ήδη στο παρελθόν μετά το τρομοκρατικό πλήγμα της 11 Σεπτεμβρίου. Νομίζω όμως ότι σε σχέση με αυτή την κατάσταση είναι πρόορη η φάση αυτή να κάνουμε μια συνολική αξιολόγηση και είναι <clears throat> καλύτερο να αποφύγουμε μια ε, αίσθηση πανικού. Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό τώρα πιστεύουμε είναι να αντιμετωπίσουμε τις ζημιές και να προσπαθήσουμε να δούμε τι μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη βέβαια ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Το ότι 1% σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάθεσή της. Το 99% είναι στη διάθεση των κρατών μελών. Είναι άδικο όλα τα προβλήματα να τα φορτωνόμαστε εμείς όταν δεν έχουμε εμείς όλα τα μέσα για την αντιμετώπιση τους. Παρακαλώ, κύριος Μπόρις. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 εσείς κάνετε λόγο για την αύξηση της ανεργίας και την επικέντρωση στην καταπολέμηση της ανεργίας ώστε να επικεντρωθούμε στην κατάρτιση, στην εκπαίδευση, ώστε να βελτιωθεί η εκπαίδευση και η κατάρτιση των Ευρωπαίων πολιτών. Θα ήθελα να σα ρωτήσω το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τα ταμεία για την έρευνα και ανάπτυξη θα διατηρηθούν στο μέλλον μέσα στο πλαίσιο του κοινοτικού προπολογισμού, διότι είναι τα κλειδιά για την καινοτομία και την καινοτόμο δράση και για μεγαλύτερη απασχόληση. Και επίση πιστεύω ότι θα έπρεπε να επικεντρωθούμε στην επένδυση, σε επενδύσει στι ε, ε, μακροοικονομικές δυνατότητες δράσης ε, στις μικροεπιχειρήσεις ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις δυνατότητες τους. Όπως γνωρίζετε στη στατική 2020 προτείνουμε ένα από τους στόχους που έχουμε συμπεριλάβει την κατάσταση και εκπαίδευση την δυνατότητα να καταπολεμήσουμε το να εγκαταλείπουν οι νέοι τα σχολεία χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών τους σε αυτά και πρέπει να το δούμε το θέμα αυτό της ε, εκπαίδευσης και της παιδιάς Γι' αυτό προσπαθούμε σε όλα τα κράτη-μέλη να ε, υπάρξει, να πείσουμε τα κράτη-μέλη να ενστερνιστούν αυτό το στόχο. Τώρα, για την κινητοποίηση των κονδυλίων, με κάποια από αυτά τα κονδύλια θα προέρχονται από τα κράτη-μέλη, κάποια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να συζητήσουμε τι δημοσιονομικέ προοπτικέ. Δεν έχει γίνει ακόμα αυτό. Κάποια δράση πρέπει να αναλυφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε τι δράσει ε, των ε, εθνικών κυβερνήσεων. Και στο κοινωνικό ταμείο υπάρχουν ήδη δράσει που προβλέπονται για νέους, για την μαθητεία και την κατάρτιση για αυτούς. Αυτό είναι ένας από τους τομείς δράσης. Τώρα, σίγουρα μπορεί το κοινωνικό ταμείο να εμπλακεί. Πρέπει να έχουμε αρκετά υψηλό επίπεδο φιλοδοξιών για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά τα ευρωπαϊκά μέσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η κυρία ε, Πρόεδρε, πληροφορηθήκαμε από τα μέσα ενημέρωσης ότι θα κλείσει η αυτοκινητοβιομηχανία Opel στην Αμβέρσα. Ένα από τα πολλά παραδείγματα για την απώλεια θέσεων απασχόλησης. Στην επόμενη Πέμπτη η, τα ευρωπαϊκά συνδικάτα θα κάνουν μια πανευρωπαϊκή διαδήλωση γι' αυτό απέτησή τους είναι η διασφάλιση της έδρας στην Ευρώπη των επιχειρήσεων και η διασφάλιση θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη από βράση αυτών των επιχειρήσεων. Θέλουν πλήρη απασχόληση και θέλουν η ευρωπαϊκή πολιτική με σθένος να ενεργοποιηθεί και να δράσει. Απαιτούν και αναμένουν συγκεκριμένες απαντήσεις σήμερα και όχι κάποτε στο μέλλον. <clears throat> Δεν είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά. Είπατε, γιατί αναφέρατε τις ε, ε, κατευθυντήριες γραμμές, τις οδηγίες και το έγγραφο θέσεων ε, Ευρώπη 2020. Αυτά δεν είναι αρκετά χειροπιαστά όμω. Τι θα κάνετε χειροπιαστά ώστε ένα στρατηγικά σημαντικό τομέα όπω η αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη να μπορέσει να υποστηριχθεί. Ποιο ρόλο διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να είναι βιώσιμο ο τομέα των αυτοκινητοβιομηχανιών στο μέλλον και να διασφαλιστεί στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Μπαρόζο, οι οδηγίε για την απασχόληση, οι κατευθυντήριε γραμμέ για την απασχόληση φυσικά επικεντρώνται στην συνολική οικονομική ανάπτυξη. Όμω η συνιστόσα τη απασχόληση πρέπει να τονωθεί και έχουμε την, αύξηση, την αυξημένη συμμετοχή στην αγορά εργασία αναπτύσσοντα καταρτισμένου εργαζόμενου την διαβίου εκπαίδευση και κατάρτιση, βελτίωση των συστημάτων παιδεία και εκπαίδευση και βελτιώνοντα τι δυνατότητε ε, επαγγελματική ανάπτυξη, καταπολέμησης τη φτώχεια και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτέ είναι οι γενικέ κατευθυντήριε γραμμέ που πρέπει να τύχουν συνέχεια και να ολοκληρωθούν από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τι εθνικέ κυβερνήσει. Αληθεύει ότι δεν υπάρχει μαγική ράβδο εδώ, δεν υπάρχει μαγική λύση για την καταπολέμηση τη ανεργία στην Ευρώπη. Πρέπει να, συνολικά πολλά μέτρα να μπορέσουν να λειτουργήσουν υπέρ της ανάπτυξης, υπέρ του ε, Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, υπέρ της ισορροπίας των αγορών, υπέρ τη της εσωτερικής αγοράς. Έτσι μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Όσον αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία, φυσικά γνωρίζαμε ότι υπήρχε πλεονάζον δυναμικό, όχι μόνο στην ε, Ευρώπη αλλά και αλλού. Παρακολουθούμε του σύνεγγυ στα τεκτενόμενα και παρακολουθούμε και με τα συνδικάτα τι δράσει του για να πετύχουμε αυτού του στόχου. Η ε, κυρία Χάνου Τάκουλα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τάκουλα, φυσικά. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Μάλιστα. Κατανόησα ότι ήταν λάθος σας. Φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Είμαι άντρας και στοχεύω να παραμείνω άντρας. Τώρα για την ερώτησή μου. Αγαπητέ Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υψηλή απασχο... ανεργία και κοινωνικός αποκλεισμός, μεγάλο πρόβλημα. 20% των νέων είναι άνεργοι και πολλοί μένουν στο περιθώριο. Πάρα πολλά από αυτά τα άτομα που είναι άνεργα είναι πάνω από 50 ετών και σε πολλά κράτη-μέλη γίνεται λόγος ότι θα έπρεπε να μπορέσουν να αυξηθεί το όριο στο οποίο, μέχρι το οποίο εργάζονται και μετά συνταξιοδοτούνται. Και υπάρχουν εδώ νομίζω αντιφάσεις σε σχέση με την κατάσταση και τα μέτρα που θέλουμε να λάβουμε. Αν θέλουμε να παρατείνουμε τον, εργάσιμο, τον, τον, τον βίο των όσων εργάζονται, γιατί τότε δεν δίνουμε τη δυνατότητα σε νέους να εργάζονται και αυτοί παραμένουν άνεργοι ποια είναι η πραγματική ευρωπαϊκή στρατηγική. Δεν μπορούμε αυτή τη στρατηγική να τη συνδυάσουμε για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Όλοι συμφωνούμε ότι οι νέοι, καταρτισμένοι, καλά καταρτισμένοι νέοι, θα πρέπει να μπορούν να βρουν μια θέση απασχόλησης ώστε να μην αποκλείονται από την κοινωνία μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα δώσει πρόσθετη αξία στην κοινωνία. Ευχαριστώ για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί σε αυτόν τον αγώνα. Ένα πράγμα είναι βέβαιο. Χρειαζόμαστε περισσότερου που θα εργάζονται, θα εργάζονται περισσότερο και επί μακρότερο χρονικό διάστημα και θα είναι και πιο παραγωγικοί. Δεν υπάρχει εδώ λοιπόν αντίφαση στο να έχουμε μεγαλύτερη, ε, ε, μακρότερο χρόνο εργασίας ε, όσον αφορά την ηλικία των όσων θα εργάζονται προτού συνταξιοδοτηθούν και μεταξύ των στόχων αυτών και τη εργασία του. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν πάνω από 500.000 ε, θέσεις ε, διαθέσιμες απασχόλησης. Ε. Και αυτό εδώ πρέπει να μας κάνει να δούμε το πώς θα μπορέσει η ζήτηση και η προσφορά να συγκλίνουν. Πολλά μπορούν να γίνουν. Πιστεύω ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι ένας τρόπος για να συνεισφέρουμε. Θέλω να υπογραμμίσω ότι κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης <clears throat> τα κράτη-μέλη σε σχέση με την παραδοσιακή πολιτική δεν ε, περίμεναν να ε, αποχωρήσουν από το χώρο εργασίας, από την εργασία τους ε, οι όσοι εργαζόντουσαν για να βρουν οι νέοι θέση εργασίας. Είναι σημαντικό αυτό όμως γιατί για να παραμείνει η Ευρώπη ανταγωνιστική πρέπει να αυξήσουμε τα όρια ηλικία και το όριο μέχρι το, οποίο, το οποίο εργάζονται οι εργαζόμενοι. Ευχαριστώ. Η κυρία Σιλιάσκα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε, Πρόεδρε Μπαρόζο, στο σημερινό σας λόγο αναφέρατε και είπατε ότι πρωταρχική προτεραιότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής όσον αφορά την απασχόληση είναι να βοηθήσετε εκείνους που τελειώνουν τα σχολεία τους ε, να μπορούν να περνάνε στην ε, αγορά εργασίας και να βρίσκουν απασχόληση. Έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό ανεργία, 40% στην Ισπανία, 20% ανεργία στον πληθυσμό και αυξάνεται αυτό το ποσοστό. Φαίνεται ότι στην Πολωνία δεν υπάρχει συμβατότητα σε σχέση με τα όσα μαθαίνουν οι νέοι όταν έρχεται η ώρα να βρουν μια θέση απασχόλησης. Σε τι οφείλεται αυτή η κατάσταση. Πώς αξιολογείται τις επιδόσεις του προγράμματος Λεωνάντο Νταβίντσι. Προετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νέες δράσεις και αν ναι τότε ποιε είναι αυτές για να μπορέσει να βοηθηθεί η απασχολησιμότητα των νέων. Τι είναι αυτό το οποίο έχετε να προσφέρετε και μπορείτε να κάνετε για τους νέους στην Ευρώπη κύριε Μπαρόζο. Η ανεργία των νέων είναι το πιο δραματικό πρόβλημα στην ε, Ευρώπη σήμερα. Είναι πάνω από 20% και γι' αυτό προαναγγείλαμε τρει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Η κινητικότητα των νέων, η ε, αποτελεσματική δράση σε σχέση με ε, την εργασία, η απασχολησιμότητα των νέων δίνει τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε τα προβλήματα αυτά και οι θέσει απασχόληση να μπορούν να δίνουν δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε τι ικανότητε αυτών των νέων. Θέλω λοιπόν αυτό να ληφθεί υπόψη. Η ε, πολιτική, η στρατηγική για το 2020 πρέπει να δούμε ότι θα απαιτεί 16 εκατομμύρια περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Και εδώ έχουμε προβλέψει μεταξύ 2007-2013 να δώσουμε ε, τα αναγκαία κονδυλία για να υπάρχει η προσαρμογή των μέτρων εκείνων που θα υιοθετηθούν. Πολλά μπορούν να γίνουν για την υιοθέτηση αυτών των ε, μέτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη για να καταπολεμηθεί το πρόβλημα της ανεργίας των νέων. Η κυρία Ελίζαμπετ Σρόιτερ παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε Μπαρόζο, πρέπει να διαφωνήσω μαζί σας. Λυπούμε, είπατε ότι μέτρα για το πράσινο δυναμικό πρέπει να εκμεταλλευτούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 2020 η στρατηγική μας κατοχυρώνονται αυτά τα μέτρα. Δεν αληθεύει αυτό. Αυτό το στοιχείο το ξεχάσατε στη στρατηγική σας και δεν έχει συμπεριληφθεί. Και διαρωτώ με γιατί. Γιατί έγινε αυτό. Διότι είναι προ... και πρόδειλο ότι αν θέλουμε να πετύχουμε μεγαλύτερη απασχολησιμότητα, μεγαλύτερη απασχόληση, το πρασίνισμα της οικονομίας δίνει τη δυνατότητα να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί απουσιάζει αυτό το στοιχείο στη στην στρατηγική του 2020 και τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε η, αϊφόρα διάσταση σε σχέση με το πρασίνισμα της οικονομίας και των δράσεων να τονωθεί περισσότερο. Θα πρέπει αυτό να γίνει από πλευρά σας. Εδώ επειδή είναι μια μεγάλη ευκαιρία, εσείς τι κάνετε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πετύχετε αυτούς τους στόχους. Ευχαριστώ. Πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ξεκίνησε το πακέτο για τις κλιματικές αλλαγές και τα ενεργειακά θέματα και ότι είδαμε ότι υπάρχει μεγάλο δυναμικό σε κάποιους τομείς για το από το πρασίνισμα της οικονομίας και αυτό σίγουρα είναι μια προτεραιότητα για το μέλλον και είναι σίγουρα μία από, ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους της στρατηγικής του 2020. Εντάξαμε στο επίκεντρο της στρατηγικής για το 2020 το κλίμα, τις κλιματικές αλλαγές, την προστασία του κλίματος και τα ενεργειακά θέματα, δίνοντας προτεραιότητα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δίνοντας τη δυνατότητα με αυτούς τους στόχους να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης σε όλους τους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Βρίσκεται στο επίκεντρο ακριβώς της οικονομικής μας στρατηγικής για το μέλλον. Και αυτό είναι ένας από τους πυρήνες της πολιτικής μας για την ανάπτυξη και για την ισόρροπη ανάπτυξη, δίκαιη ανάπτυξη και αηφόρα ανάπτυξη. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Η τελευταία ερώτηση τώρα, παρακαλώ. Λίσα Γιακονσάρη, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, συζητήσαμε, κάναμε λόγο για τους νέους εδώ. Μία άλλη ομάδα όμως που αντιμετωπίζει ανεργία είναι οι γυναίκες. Ακριβώς οι γυναίκες. Τώρα που οι οικονομίες μας είναι υπερχρεωμένες και πιέζονται και κάνουν περικοπές στους προϋπολογισμούς τους στα κράτη-μέλη. Αυτές οι περικοπές στοχεύουν σε πολλούς τομείς όπως την κατάρτιση και παιδεία και όσον αφορά και την εργασία των γυναικών πλήττουν ιδιαίτερα τις γυναίκες. Θα ήθελα να μου πείτε Πρόεδρε Μπαρόζο, τι θα κάνετε ακριβώς σε εκείνα τα κράτη-μέλη όπου άσχετα από το γεγονός ότι το πρόγραμμα για τη στρατηγική του 2020 λέει ότι θα έπρεπε να έχουμε στόχους να ενδυναμώσουμε το ανθρώπινο δυναμικό, την υγεία, την περίθαλψη. Υπάρχουν περικοπές όμως και από τα κράτη-μέλη στόχος τους είναι να περικόπτουν διαρκώς κονδύλια, να περικόπτουν διαρκώς. Τι θα κάνετε εσείς σε σχέση με αυτή την κατάσταση και αυτά τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Uh, σας ευχαριστώ για τις γυναίκες. 9,3% το Φεβρουάριο του 2010 σε σχέση με τον 9,8% ε, των ανδρών. Χαμηλότερο ποσοστό από των ανδρών δηλαδή. Αλλά αληθεύει αυτό που είπατε ότι δημιουργεί μεγάλες ανησυχίες ε, η ανεργία των γυναικών. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις μελλοντικές προοπτικές. Κάποιοι τομείς ε, θα, έχουν, θα πληγούν περισσότερο σε σχέση με κάποιες περικοπές διότι εδώ έχουμε το θέμα θέμα της απασχόλησης των γυναικών κατά κύριο λόγο σε αυτούς τους τομείς. Πρέπει να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τις πολιτικές τους ως προς τις επιπτώσεις τους, να μην είναι οι γυναίκες τα θύματα, διότι πιστεύουμε ότι ο στόχος όσον αφορά την απασχόληση και το έχουμε συζητήσει με τα κράτη-μέλη και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι στόχοι, το ποσοστό δηλαδή ε, όσον αφορά την ε, ε, ε, ανάπτυξη και την απασχόληση πρέπει να επιτευχθεί όσον αφορά και τους άνδρες και τις γυναίκες. Σε κάποια κράτη-μέλη έχουμε μεγάλο δυναμικό. Έχουμε κάποια κράτη-μέλη όπου είναι πολύ χαμηλότερο το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών σε σχέση με εκείνο των ανδρών. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις απαντήσεις σας. Προσβλέπουμε στην συνεργασία σας και την παρουσία σας σε επόμενη περίοδο χρόνου ερωτήσεων εδώ στην Ευρωβουλή σας ευχαριστώ. Θα συναντηθούμε πάλι τον επόμενο μήνα στον χρόνο ερωτήσεων με τον κύριο Πρόεδρο Μπαρόζο. Σας ευχαριστούμε πολύ.